Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα πάγιο μέλημά μας. Ε, προχωρώ τώρα στα συνοπτικά πρακτικά ε, που διανεμήθηκαν τις 12 Νοεμβρίου και τα κείμενα που εγκρίθηκαν τότε. Έχετε λάβει τα συνοπτικά πρακτικά, δεν ξέρω αν έχετε σχόλια και παρατηρήσεις, ερωτώ. Θέλει κανείς να ε, λάβει το λόγο σχετικά με τα συνοπτικά πρακτικά της 12 Νοεμβρίου, όχι. Εγκρίνονται λοιπόν. Επόμενο θέμα. Οι αρμόδιες τσεχικές ε, αρχές